επισκεπτών της υποτροφίας Ζαχάροφ που δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 14 ε, υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστές από διάφορες χώρες έχουν αυτή την υποτροφία και είναι από τη Λευκορωσία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Γουατεμάλα, Ιράν, Ιορδανία, Καζακστάν κλπ. Παρακολουθούν ένα εντατικό σεμινάριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύο εβδομάδων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και ε,